ΓΚΟΕ και την ΙΕΝΕΦ e έτοιμα για την ΙΤΡΕ, ε, ούτω ώστε να αρχίσουν οι διοργανικέ διαπραγματεύσει όσον αφορά την έκθεση για του κοινού ε, κανόνε εσωτερική αγορά για το φυσικό αέριο και εν προκειμένου εισηγητή ο κ. Μπούζεκ θα γίνουν αύριο οι σχετικέ ψηφοφορίε όσον αφορά την απόφαση, ούτω ώστε να αρχίσουν οι διαπραγματεύσει από την ΤΡΑΝ και την ΕΜΠΛ. Ε, δεν έχω έτοιμα σε σχέση με ψηφοφορία. Οπότε μπορούν αυτές οι επιτροπές να αρχίσουν διαπραγματεύσεις και επίσης σας ανακοινώνω ότι ο κύριος Σοπράντ δεν είναι πλέον ε, στους μη εγγεγραμμένους και προσεχώρησε στην ομάδα EFDD κάτι το